Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά αυτά. Περάμε σε ανακοινώσει του Πρόεδρου. Δύο βουλευτέ δήλωσαν ότι κρατούνται <coughs> από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρια Νταϊάννα Νταγιάννα Βόλη. Από Φεβρουαρίου 2012 εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βόλη για την πολυετή επικοδομητική και επιτυχή εργασία τη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, ο κ. Πρόεδρο Αστερόσα, ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα Φεβρουαρίου <clears throat> καταθέτει την εντολή του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τα συγχαρητήρια εσύ και για τον ίδιο. Ελπίζω ότι θα έρθει σε λίγο και μπορείς να το ευχαριστήσω και προσωπικά. Το σώμα το σημειώνει και η βάση του άρθρου 4, παραγραφή 1 και 3 του κανονισμού σημειώνει ότι οι έντρες αυτές χειρεύουν από τις ημερομηνίες που προανέφερα. Ο κ. Βιλέιταλα μου ανακοίνωσε ότι ορίστηκε μέρο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Το σημειώνει το Κοινοβούλιο αυτό και βάσει το άρθρο 4, παραγράφη 1 και 4 του κανονισμού σημειώνει την χειρία τη έδρας του κ. Βίτα Ιταλά από την 1η Μαρτίου 2012. Θα ήθελα επίση να σα ανακοινώσω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων